Ο κύριος Μπρίς Ορτεφέ υπέβαλε στην, στο Προεδρείο αίτημα υπεράσπισης της βουλευτικής του ασυλίας και των προνομίων του στα πλαίσια δικαστικής εξέτασης που έχει ξεκινήσει στο Παρίσι. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό το αίτημα προωθείται προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις στην σύσταση της απόφασης της